υποστηρίξει για να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί από την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πέρα στη συζήτηση θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. έκθεση της κυρίας Γουόλη σχετικά με τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε υποθέσεις του αστικού, εμπορικού και οικογενειακού δικαίου. Η εισηγήτρια έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε. Εναλλακτικέ ε, δυνατότητες επίλυσης διαφορών ουσιαστικά όσον αφορά το αστικό δίκαιο και εμπορικό δίκαιο αλλά επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε θέματα καταναλωτών αυτό για το οποίο κάνουμε λόγο είναι να υπάρχει πρόσβαση στην δικαιοσύνη και ρύθμιση θεμάτων και κάνοντας αυτό να βρούμε ένα τρόπο να ενθαρρύνουμε διασυνοριακές συναλλαγές διότι αυτή τη στιγμή επί πολλά χρόνια υπάρχουν φόβοι όσον αφορά την επιβολή δικαιωμάτων. Οι παραδοσιακές διεργασίες δικαιοσύνης είναι περίπλοκες, ε, βραδίες ε, και δαπανηρές. Ταυτόχρονα όμως σε μια εποχή που θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις ε, διασυνοριακές συναλλαγές πρέπει να βρούμε, ας το αποκαλέσουμε έτσι, ένα νέο πολιτισμό αστικού δικαίου και δικαιοσύνης, διαφορετικό του, του παλαιού, που θα είναι πιο φθηνές οι διαδικασίες, λιγότερο δαπανηρές και ταχύτερες για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Επί πολλά χρόνια υπήρχε ένα χαλαρό δίκτυο παρόχων που συντονιζόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το EGNet και το FinNet ως δίκτυα. Ήταν επιτυχή κατά έναν τρόπο, αλλά δεν επαρκούν από την άλλη πλευρά δεν δίνουν λύσεις στα ζητήματα που θα έχουν και τα ερωτήματα που θα έχουν οι περισσότεροι πολίτες όταν θα επιθυμούν να απονεμηθεί δικαιοσύνη που θα γνωρίζουν ε, κάποια πράγματα δεν θα ξέρουν τι θα γίνεται με το EDR. Πρέπει τα συστήματα αυτά να διαχυθούν και να διαδοθούν ώστε να τα γνωρίζουν οι πολίτες. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο συνολικό σύστημα όπου κάθε καταναλωτής θα μπορεί να καταλήγει σε ένα EDR σύστημα για την επίλυση διαφορών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συστήματα που υφίστανται θα είναι καλής υψηλής αναβαθμισμένης ποιότητας, ότι θα υπάρχει κατάρτιση για αυτούς που εμπλέκονται και παρέχουν υπηρεσίες στο ADR και θα υπάρχει μια αμερόληπτη εποπτεία. Αυτή λοιπόν είναι η κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να πορευθούμε. Όχι απλώς ένα ADR, θέλουμε επίσης, επίσης και το ODR, Online Dispute Resolution, στο διαδίκτυο δηλαδή δυνατότητα επίλυσης διαφορών. Σε διασυνοριακές συναλλαγές πρέπει να υπάρχει online, διαδικτυακά η δυνατότητα, ηλεκτρονικά να βρίσκεται ε, λύση σε αυτές τις ε, ε, τριβές. Όμως από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να υπάρχει μία και μόνη δυνατότητα. Πρέπει να υπάρχει κοινή δυνατότητα δράσης με άλλα κοινοτικά μέσα. Η πρόταση για το συμβατικό δίκαιο, το οποίο το αποκαλούμε sales law, για τη συλλογική λογική ρύθμιση θεμάτων. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να έχουν και μια συνιστόσα ADR. Η εναλλακτική λοιπόν δυνατότητα επίλυσης διαφορών πρέπει να κάνει λόγο για μια νέα μορφή διασυνοριακής απονομής δικαιοσύνης, αλλαγή πολιτισμού όσον αφορά την προσέγγιση αυτών των θεμάτων, αλλαγή κουλτούρας συνολικά σε ένα οικουμενικό πλαίσιο. Το πιο δύσκολο θα είναι να μπορέσουμε σε σχέση με τους καταναλωτές να παράσχουμε αυτές τις υπηρεσίες στους μικρομεσαίους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους. Πρέπει να το κάνουμε ως προτεραιότητα και προσβλέπει το Κοινοβούλιο να δει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τα τέλη του 2011. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με το Κατστιάι. Η κυρία Μετζάρος έχει το λόγο. Ο κύριος Μετζάρος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η εναλλακτική δυνατότητα επίλυσης διαφορών είναι κάτι σημαντικό. Είναι μια τεχνική δυνατότητα που ευρύτατα χρησιμοποιείται και έχει τεράστια σημασία όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις. Η νομική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και η κυρία Γόλη συνέταξε την έκθεσή της εκκινώντας από το σκεπτικό ότι τα στοιχεία, οι αριθμοί δείχνουν ότι μία πλούστευση, ένα πιο διάφανο πλαίσιο για την επίλυση διαφορών στην Ευρώπη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν απαραίτητο είναι επιτακτική ανάγκη. Τα κράτη-μέλη και οι εξειδικευμένες ενώσεις και σύλλογοι να μπορέσουν με αποτελεσματικό τρόπο να συνεργαστούν. Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τις πιο διαφορετικές δυνατότητες του ADR μπορεί να δώσει την δυνατότητα εξοικονόμησης δαπανών και κόστους για την κοινωνία μας και τους πολίτες. Επιπρόσθετα για τα ειχέγγυα, για τις εγγυήσεις, είναι έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενημερώνει για τα προτερήματα προβλήματα του ADR συνολικά. Ευχαριστούμε. Ρέιτοβα στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Πάντα υποστήριζα το ADR. Έχω όμως μια σημαντική επιφύλαξη <clears throat> Αυτό είναι η συμπερίληψη οικογενειακών θεμάτων, οικογενειακού δικαίου ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό, αυτός ο τομέας εντάσσεται στην νομοθεσία των κρατών μελών και επικυριαρχία των κρατών μελών. Περίπλοκες ε, οικογενειακές υποθέσεις που αφορούν και τα παιδιά πρέπει να κρίνονται από εξειδικευμένους, καλά καταρτισμένους δικαστές και δεν θα πρέπει να παρισφρέει και να αναμειγνύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζουμε όμως ε, τα συστήματα ADR σε άλλα θέματα, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα καταναλωτών και εμπορίου, επειδή είναι λιγότερο δαπανηρά, ταχύτερα, πιο αποτελεσματικά. Αυτά τα συστήματα πρέπει να αναπτυχθούν ω συστήματα που εξαρτώνται από το διαδίκτυο και πρέπει να ενταχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επωφελή για επιχειρήσει και να συμμορφώνονται με την αρχή τη αμεροληψία, διαφάνεια, δικαιοσύνη. Πολλέ φορέ επεσήμανα ότι θα πρέπει η πείρα μα σε σχέση με, το, με τα ADR να χρησιμοποιείται όσον αφορά τα ηλεκτρονικά μας μέσα. Ολοκληρώνω. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση ώστε να μπορέσουν να διαδοθούν στην Τσεχία αυτά τα... Και κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γουόλης για την έκθεση της στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η πρόσβαση των καταναλωτών και των ΜΜΕ στις διαδικασίες εναλλακτική επίλυσης διαφορών είναι ουσιαστικές για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς διότι επιλύουν γρήγορα τις διαφορές και με μικρότερο κόστος. Τα εμπορικά δικαστήρια και τα ειρηνοδικεία λειτουργούν στα κράτη-μέλη αλλά λύνουν τα προβλήματα μόνο σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται εναρμόνιση σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Δύσκολα όμως μπορούν να λυθούν διαφωνίες όταν έχουμε, όταν έχουμε τέτοια διαφορετικά δικονομικά συστήματα. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να έχουμε μία εναρμόνιση όλων αυτών των κανόνων για να λύνονται τέτοιου είδους διεθνείς διαφωνίες. Ευχαριστώ. Εκτίμησα ιδιαίτερα στην έκθεση Wallis το γεγονός ότι θέλει μία γενική ατζέντα για την ανάπτυξη εγκάρσια που θα λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα αστικού, εμπορικού και οικογενειακού δικαίου. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι διαφορές σε επίπεδο οικογενειακού δικαίου και αυτό κυρίως μετά από διαζύγια σε διευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε διαφωνίες μεταξύ πολιτών διαφορετικής υπηκότητας που εμπίπτουν κυρίως στην πλάτη των παιδιών. Το να μπορούμε να έχουμε εμεί έναν ουδέτερο οργανισμό στον οποίο κανείς μπορεί να προσφεύγει, μπορεί να οδηγεί στο να παρουσιάζουμε λύσεις ισορροπημένες με ομολογοποίηση προς τον δικαστή γίνεται σεβαστή ημένη η επικουρικότητα και στο πλαίσιο των κανονισμού 2005 για την οικογενειακή ευθύνη και περιφρουρούμε και τη διασυνοριακή προστασία των ανήλικων. Εύχομαι λοιπόν η Κομισιόν να δει και αυτή την πτυχή προς την κατεύθυνση των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Κυρία Φλασίκοβα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η προσπελασιμότητα στη δικαιοσύνη και τις υπηρεσίες της είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα και η εναλλακτική επίλυση διαφορών και η αναζήτηση λύσεων είναι εκείνη που μπορεί να επιλύσει προβλήματα των δύο πλευρών χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια. Δίνει επίσης την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί κάποιος τρίτος εκτός δικαστηρίων ως διαμεσολαβητής. Υπάρχει εδώ δηλαδή με λιγότερες δαπάνες η δυνατότητα ρύθμισης διαφορών έναντι της προσφυγής στα δικαστήρια. Είναι κρίμα ότι η πληροφόρηση στα κράτη-μέλη για τις δυνατότητες του ADR είναι περιορισμένες οι δυνατότητες πληροφόρησης στα κράτη-μέλη, διότι λίγοι γνωρίζουν πού πρέπει και πώς πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ίσως για αυτούς τους λόγους πρέπει να ενημερώσουμε, να πληροφορήσουμε περισσότερο τους πολίτες για την ύπαρξη και διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών. Είναι μια δυνατότητα να αποφύγουμε ε, με τοπική αντιπαράθεση και σύγκρουση και είναι η δυνατότητα που παρέχεται να εξευρεθεί λύση ικανοποιητική για αμφότερες τις πλευρές. Όμως θα πρέπει να είναι ισορροπημένη η πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία ώστε να απονέμεται δικαιοσύνη σε αμφότερες πλευρές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Υποστηρίζω την ιδέα του να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια κοινά σημεία επαφής και συνεννόησης. Είναι καλό όμως να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο για την εναλλακτική επίλυση διαφορών σε θέματα αστικού δικαίου αλλά και στα θέματα οικογενειακού δικαίου για να πλουστευτεί η ζωή των πολιτών. Να βρούμε μια εξοδικαστική δυνατότητα επίλυσης που, έχει, ε, που είναι υποφελές για όλους. Η οικογένεια όπως αναφέρεται στον τίτλο της έκθεσης όμως δεν βρίσκεται, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εκείνων όπου θα μπορούσε να γίνει χρήση αυτών των δυνατοτήτων. Η κυρία Ρότοβα το ανέφερε. Δεν μπορούμε ισοπεδωτικά να εφαρμόσουμε μία αρχή σε όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν προβλήματα εδώ τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη προβλήματα και που μπορούν να δημιουργηθούν κιόλα αν προσπαθήσουμε να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση για θέματα ε, διαζυγίου για παράδειγμα και πρέπει να τα δούμε αυτά. Πάσκα. Κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η εναλλακτική επίλυση διαφορών εξοδικαστικά αλλά και για θέματα οικογενειακά θα, μπορούσαν, θα μπορούσε να συνεισφέρει για την ειρηνική επίλυση διαφορών και έτσι θα πρέπει να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τις ε, δυνατότητες που προσφέρει αυτή η ρύθμιση νομοθετικά. Ιδιαίτερα η ρήτρα που προβλέπει διαδικασίες ε, για τις, ε, την ανάκτηση μικροποσών όσον αφορά εμπορικά ζητήματα. Είναι μια πολύ καλή βάση για εναλλακτική αναζήτηση επίλυσης διαφορών σε διασυνοριακές συναλλαγές. Συμφωνώ με την άποψη ότι η ενημέρωση των πολιτών μπορεί να βοηθήσει στη διάδοση και διάχυση αυτών των δυνατοτήτων και της αύξησης ε, της εναλλακτική επίλυσης διαφορών. Επίσης η εξοδικαστική δυνατότητα ρύθμισης διαφορών θα μπορούσε να μειώσει και την ψυχολογική πίεση και το άγχος όσον αφορά οικογένειες και μέλη οικογενειών αν δει κανείς και συγκρίνει με τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται από πλευράς δικαστικής προσφυγής και αυτό θα ήταν υποφελές. Ευχαριστώ. Ehm, η Επίτροπος, κυρία Ρέντινγκ. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η Επιτροπή σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ε, σχετικά με ε, την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Να καλωσορίζουμε τις ε, προτάσεις που κάνετε σχετικά με την νομοθετική πρόταση για τις διαφορές των καταναλωτών. Η δήλωση της Κρακοβίας που ενέκρινε το Φόρουμ της Νέας Αγοράς νωρίτερα επανέλαβε τις ίδιες αρχές. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι μία από τις 12 προτάσεις της πράξης για την ενία αγορά. Ο συνάδελφός μου, Επίτροπος Νταλή, θα καταθέσει δύο νομοθετικές προτάσεις. Βλέπετε να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 31η Οκτωβρίου μια οδηγία πλαίσιο για, ε, τις, για τις εναλλακτικές ε, επιλύσεις διαφορών και μια οδηγία για την ε, γραμμική επίλυση διαφορών με πρόβλεψη ε, ούτως, ώστε οι καταναλωτές για οποιαδήποτε αντιδικία να έχουν πρόσβαση. Θα έχουμε δικτυακή πύλη επίσης για τις επιγραμμικές ε, συναλλαγές ανάμεσα στους καταναλωτές και τους εμπορευομένους. Ε, αυτές οι προτάσεις θα είναι τα πρώτα τουβλάκια αν θέλετε στην οικοδόμηση ενός νέου συστήματος εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών. Η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα business to business, δηλαδή σχέσεις επίλυση διαφορών ανάμεσα στι επιχειρήσεις, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κάτι διάρκεια των διαβουλεύσεων για τις αντιδικίες ανάμεσα στι επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Οι εμπλεκόμενοι φορείς αφέστατα εξέφρασαν προτίμηση για ε, διαφορετικού τύπου τύπου εργαλεία, ε, δηλαδή για να εφαρμοστούν διαφορετικού τύπου εργαλεία και μέσα για τις αντιδικίες ε, ε, ανάμεσα στις επιχειρήσεις B2B και εξετάζουμε το ενδεχόμενο επιδιαιτησίας κυρίως στις διασυνοριακές αντιδικίες από επιχείρηση σε επιχείρηση. Είμαστε ακόμη σε πρόωρο στάδιο, συλλέγουμε πληροφορίες και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορέσουν να παρεμποδίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα δραστηριότητα κυρίως των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου καλωσορίζουμε όλες ε, τις ε, προτάσεις κατά την επεξεργασία του ζητήματος και ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη πρόταση επίσης για την οδηγία περί επιδιαιτησίας ε, κυρίως στον τομέα οικογενειακού δικαίου, όταν μιλάμε για τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, ε, δηλαδή όταν δεν καταφέρνουν να επιλύσουν τη διαφορά σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, θέλουμε να υπάρχει μια αναλλακτική επίλυση διαφορών, ώστε να μην μπουν σε χρονοβόρες ε, δικαστικές διαδικασίες. Από την 21η Μαΐου του 2011 σε όλες τις χώρες εκτός από τη Δανία εφαρμόζεται αυτή η οδηγία για αστικά εμπορικά ζητήματα, ζητήματα οικογενειακού δικαίου καθώς και αντιδικές ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν ε, οι αντιδικοί δεν μπορούν να αποφασίσουν ε, τα, ε, για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους βάση του εφαρμοστείου οικείου δικαίου. Ευχαριστούμε το κοινό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του σχετικά με τι βασικέ διατάξει ω προ την οδηγία επιδιαιτησία ε, που θα έπρεπε να εφαρμοστούν και σε άλλου μηχανισμού ε, εναλλακτική επίλυση ε, διαφορών. Μιλάμε για την παραγραφή, για την εφαρμοστικότητα των νομοθετικών διατάξεων κτλ. κτλ. Δηλαδή για τα, όλα τα κοινά πρότυπα που θα διέπουν την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Μετά την έναρξη των διαδικασιών επί παραβάση κατά εννέα κρατών μελών τον Ιούλιο λόγω της αργοπορίας στη μεταφορά της οδηγίας στην Εθνική Νομοθεσία. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι 21 κράτη-μέλη έχουν κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας στην επικράτειά τους και παρακολουθώ εκ του σύνεκης εξελίξεις και στα λοιπά κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Πέρα τη συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. Έκθεση του κυρίου